Άρχεται η συνεδρίαση. Καλημέρα σε όλους και όλες. Αδελφοί, αγαπητοί συνάδελφοι. Ναι, παρακαλώ. Ένα ερώτημα μονάχα σε σχέση με την ημερήσια διάταξη, κύριε Πρόεδρε. Στις 12 είναι προσκεκλημένος ο Φίλιππος της Φουρβονίας για να λάβει το λόγο ενώπιον της ε, Ολομέλες εκφράζω την απόρριψή μου, γιατί αυτό το κοινοβούλιο πρέπει να εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία και επομένω θα πρέπει να έχει κλειστέ τι πόρτε του στου επικεφαλεί κρατών οι οποίοι δεν έχουν εκλεγεί δημοκρατικά και αυτό δεν ισχύει για τον βασιλιά τη Ισπανία. Γι' αυτό ζητούμε από την Ολομέλεια να μην επιτρέψει ένα επικεφαλή κράτου ο οποίο δεν έχει δημοκρατική νομιμοποίηση να λάβει τον λόγο ενώπιον τη Ολομέλεια. Ευχαριστώ. Εγώ δεν βλέπω καμία παραβίαση των δημοκρατικών παραδόσεων, ε, κυρία Βουλευτή, να υπάρχουν προσκεκλημένοι. Περνάμε στο πρώτο σημείο τη ημέρα τη διάταξη. Είναι η δήλωση τη ΥΠΑ του εκπροσώπου και αντιπρόεδρου τη ε, Κομισιόν, υπεύθυνη για εξωτερική πολιτική και θέματα ασφαλεία, σε σχέση με την αεροπορική επιδρομή εναντίον ενό νοσοκομείου στο Αφ... Κούντου του Αφγανιστάν. Δεν θα υπάρξει διαδικασία eye για αυτήν την συζήτηση, ούτε θα γίνουν δεκτέ μπλε κάρτε. Ξεκινούμε με την δήλωση από, τον, από την Αντιπρόεδρο, την οποία εκπροσωπεί ο κύριος Στυλιανίδη.